επίπεδο της σταθερότητας της χώρας. Εδώ λοιπόν η απάντηση που ήθελα να δώσω εκ μέρους της κυρίας Άστον και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Μπαρνιέ. Η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί εδώ. Και επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τον διορισμό των Προέδρων των διαφόρων ευρωπαϊκών εποπτικών οργάνων. Και θα ήθελα να καλέσω την κυρία ε, Γκέρι καταρχήν. Εξ Συμβουλίου, κυρία Κύριε Επίτροπε, αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να σχολιάσω από πλευράς του Συμβουλίου τις διαδικασίες των θέσεων των νέων εποπτικών αρχών και των αρχών επίσης που θα πρέπει να διέπουν τις, ε, την αποστολή τους. Δεν μας έχουν δοθεί ξεκάθαρες οδηγίες στο Συμβούλιο σχετικά με τον διορισμό αυτό. Ο πρόεδρος κάθε εποπτικής αρχής διορίζεται από το Διευθυντικό Συμβούλιο και επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την δυνατότητα να φέρει αντιρρήσεις στον διορισμό αυτών των ε, υψηλών υπαλλήλων. Τώρα το Συμβούλιο λοιπόν τι ρόλο καλείται να παίξει. Το Συμβούλιο είναι συνομοθέτης και συμφώνησε με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε ο Πρόεδρος, ο Εκτελεστικός Διευθυντής και το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε διοικητικής αρχής, εποπτικής αρχής, μπορεί να λειτουργεί πλήρως ανεξάρτητα προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σταθώ ιδιαίτερα στα άρθρα 46, 49 και 62 τα μέλη του Συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου και ο εκτελεστικός διευθυντής δεν λαμβάνουν οδηγίες από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλη κυβερνήσεων κρατών μελών και δεν θα πρέπει να προσπαθήσει κανείς από αυτούς που προανέφερα να επηρεάσουν τον πρόεδρο και τον εκτελεστικό διευθυντή των εποπτικών αρχών. Ο κανονισμός προβλέπει ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν οι κανονισμοί ε, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε ο πρόεδρος και ο εκτελεστικός διευθυντής κάθε εποπτικής αρχής να επιλέγεται σύμφωνα με τις αυστηρές βάσεις των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 48 και 51 του κανονισμού. Πέραν της διαχειριστικής εμπειρίας απαραίτητης για τον εκτελεστικό διευθυντή. Απαιτείται στα κριτήρια να περιλαμβάνονται η γνώση των αγορών, η γνώση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ε, αντίστοιχη εμπειρία σε ε, ρόλους και σε θέσεις σε ρυθμιστικές αρχές, σε εποπτικές μάλλον αρχές. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και το Συμβούλιο και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν υπεύθυνε αρχές ε, για τα δημοσιονομικά να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σε αιτήσια βάση επί τη βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σαν Προεδρία δίνουμε ε, ιδιαίτερο βάρος έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να παίξουν τον ρόλο τον οποίο καλούνται να έχουν είναι απαραίτητο όλες οι προβλέψεις των κανονισμών να εφαρμοστούν με σωστό τρόπο. Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν θεματοφύλακα των συνθήκων να διασφαλίσει τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού να ορίσει αυτούς οι οποίοι θα κάνουν τις πρώτες επιλογές στα διοικητικά συμβούλια και στις θέσεις του Προέδρου κτλ. Ελπίζω λοιπόν να προχωρήσει η διαδικασία έτσι ώστε οι νέες αυτές εποπτικές αρχές να μπορέσουν να καταστούν λειτουργικές το ταχύτερο δυνατόν είναι αναπόσπαστο τμήμα της απάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ε, προκλήσεις τις οποίες θέτει η δημοσιονομική αλλά και η χρηματοπιστωτική κρίση. Και γι' αυτό θα ήθελα να έχω την πλήρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εύρυθμη λειτουργία των ε, νέων εποπτικών αρχών. Έχει μια νέα δομή πλέον λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο εποπτικών αρχών και θα πρέπει οι εποπτικές αυτές αρχές να αρχίσουν να λειτουργούν το ταχύτερο δυνατό. Εγώ ως εκπρόσωπος της ε, Προεδρίας θα προσπαθήσω να εργαστώ αρμονικά, να συνεργαστώ αρμονικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να θεωρώ πάντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν ένα πιστό εταίρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γκιόρη. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Υπουργό Γκιόρη. Ευχαριστώ τους παρόντες ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει από την 1η Ιανουαρίου στη διάθεσή της ένα νέο εποπτικό σύστημα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το σύστημα αυτό οδηγεί σε μία σε βάθος μεταρρύθμιση των αγορών και θα ε, βοηθήσει στην σταθερότητα των αγορών και θα βάλει ε, σταθερότερα θεμέλια στην ε, χρηματοπιστωτική θα έλεγα βιομηχανία τόσο σημαντική στις χώρες μας. Θα ήθελα εδώ να χαιρετήσω τον Μίζωνα ρόλο, τον οποίο παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ότι σήμερα έχουμε ένα τέτοιο υποπτικό σύστημα πιο αποτελεσματικό στον αφορά το πιστοτικό τομέα και εάν ε, για αυτό το θέμα μπορούμε να αντλήσουμε κάποια μέρα από την κρίση. Αυτό οφείλεται ω επιτοπλίστων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε αυτό το οφείλουμε. Και τώρα για να δούμε, θα πρέπει να δούμε τι τελευταίε ε, ε, φάσεις για ε, αυτές τις τρεις ευρωπαϊκές αρχές και αυτό θα γίνει ορίζοντας τον πρόεδρο και τον πρόεδρο για τον εκτελεστικό ε, διευθυντή. Αυτό θα πρέπει να γίνει με μεγάλη διαφάνεια και με, με σεβασμό τους κανονισμούς όπως αυτοί θεσπίστηκαν από τις αρχές και έτσι θα πρέπει να ορίσουμε τους, τα, τα στελέχη αυτά. Έχουμε περίπου 275 υποψηφιότητε, τι οποίε ελάβαμε όσον αφορά αυτέ τι έξι θέσει για τι οποίε σα ομίλησα. Όλε αυτέ οι υποψηφιότητε ε, εξετάστηκαν ενδελεχώς και ε, ενεπλάκησαν όλοι οι Κομισιόν, το Κοινοβούλιο επίσης ε, ε, ρωτήθηκαν και έγινε σεβαστή γνώμη οπότε και για τις επόμενες φάσεις θα προσπαθήσουμε να γίνει σωστός σχεδιασμός να υπάρχει διαφάνεια αυτή τη διαδικασία και έτσι να είναι δυνατόν η Οικονομική Επιτροπή επίσης του Κοινοβουλίου να μπορέσει να διαδραματίσει το σημαντικό της ρόλο το Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί σε σχέση με ε, μια άλλη προϋπόθεση, κάτι το οποίο απαιτείται να γίνει για αυτή την αρχή, δηλαδή αυτά τα οποία ζητείτε μπορώ να τα κατανοήσω διότι και εμείς όπως και εσείς θεωρούμε ότι ο πρόεδρος και ο εκτελεστικός διευθυντής αυτής της αρχής θα πρέπει να επιλεγεί επί τη βάση του, των προσόντων του, της ε, ε του, ε, της εμπειρίας του και για το κατά πόσον έχει γνώση του αντικειμένου αλλά και της νομοθεσίας που διέπει τις χρηματοπιστωτικές ε, αγορές. Οπότε αυτό το πνεύμα μας έχει διαπνεύσει μέχρι τώρα από τότε που υπευλήθησαν οι υποψηφιότητες. Οπότε και έτσι γίνεται και συνεχίζεται η επιλογή. Οπότε αποφασίστηκε επί τη βάση του άρθρου 68 του κανονισμού που εθέσπισε αυτήν την υποψηφιότητα ότι ο πρόεδρος και ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να υπόκεινται ή τους κανόνες για τα πρόσωπα που έχουν τέτοιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς θα υποπτεύσουμε ότι και σε σχέση με αυτό όπως και σε άλλες περιπτώσεις θα τηρηθούν οι, οι κείμενοι κανονισμοί Τώρα, όσον αφορά τους μισθούς, και αυτό σας έχει απασχολήσει, και εδώ έχουμε το ελάχιστο, το μέγιστο τέλος πάντων, το οποίο ορίζεται όσον αφορά ε, αυτά τα στελέχη, οπότε έτσι θα διερευνήσουμε τα πάντα, ούτως ώστε να υπάρχει όσο είναι μεγαλύτερη ευελιξία και για αυτόν τον τρόπο επίσης να δούμε και πώς θα υπάρξει κάποιο είδους αναθεώρηση για τη λειτουργία αυτών των αρχών όπως αυτό προβλέπεται για το τέλος του 2013. Επίσης δεν μπορώ πάνω να συμφωνήσω σε αυτό το οποίο θέλει το Κοινοβούλιο δεν εξασφαλίσει μια μεγαλύτερη ε, ισορροπία της σύνθεσης ανδρών γυναικών όσον αφορά αυτή τη, την διοίκηση αυτών των ε, υπηρεσιών οπότε και εμείς θέλουμε να ισχύει η ισότητα των ευκαιριών και αυτό ξεκινά με την διαλογή, επιλογή αυτών των υποσχετήτων που υπευλήθησαν και σε σχέση με αυτό όσον αφορά αυτή την τελευταία φάση της, ε, της επιλογής όσον αφορά τους εκτελεστικούς διευθυντές τώρα ολοκληρώνεται η διαδικασία έχουμε δύο γυναίκες οι οποίες τώρα ανταγωνίζονται για το οποίο θα καταλάβει την λόγο θέση επίσης συμφωνώ 100% με το Κοινοβούλίο και εις το εξή. Ότι δηλαδή χρειάζεται μια ισχυρή ανεξάρτητος αρχή η οποία να στερείται ή ασδήποτε παρεμβάσεις πολιτικής ή άλλης και να έχει εκκλησικό διευθυντή ούτω ώστε να είναι δυνατόν να ενεργεί αυτό και τα άλλα στελέχη με πλήρη ανεξαρτησία η ιδία, το συμφέρον τη ενώσεω. Οπότε και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αυτό το έβαλαν στο σώμα του σχετικού κανονισμού και έχουμε το άρθρο 42 και το άρθρο 46, 49 και το 52 όσον αφορά αυτά τα οποία μα υπενθύμησε και η πρόεδρο του Συμβουλίου Προεδρεύουση κυρία Γκιώρη. και οπότε και αυτόν τον τρόπο και εμείς τώρα πρόκειται 100% να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ούτως ώστε να γίνει πλήρης εφαρμογή αυτών των άρθρων. Οπότε και θα παγκρινούμε το ώστε πάσα απόφαση που να λαμβάνεται να εξυπηρετεί τα συμβούλια της ενώσεως και τώρα δούμε τα της σύνθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου. Ήδη έχουμε επισημάνει νομικά την ανάγκη και την πολιτική σημασία αυτά τα συμβούλια να απαρτίζονται από τους επικεφαλείς των αντίστοιχων αρμόδιων εθνικών αρχών. Ήδη απέστειλα τη σχετική επιστολή ώστε να διευκρινιστεί αν χρειάζεται αυτό το ζήτημα. Και ορισμένε μάλιστα από τις εθνικές αντιπροσωπείες έχουν αλλάξει ονόματα. Θα παρακολουθήσουμε από τους ε, την υπόθεση αυτή και θα δείξουμε άτεκτη στάση. Η σύνθεση θα πρέπει να είναι πλήρω συμβατή με τη δική σα βούληση, τη βούληση εν γέννη του Ευρωπαίου νομοθέτη και προσωπικώ δεσμεύονται να παρακολουθώ τουλάχιστον δύο φορέ το χρόνο τη λειτουργία με βάση το άρθρο 40 των κανονισμών που θέσπισαν αυτές τις αρχές. Και εν τέλει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, συμφωνώ με την βούληση του Κοινοβουλίου ώστε αυτές οι αρχέ να διαθέτουν τα απαραίτητα χρηματοπιστωτικά μέσα και του ανθρώπινους πόρου που απαιτούνται για την ε, επιτέλεση του έργου του κατά τρόπο απολύτω αξιόπιστη. Θα υπάρχει βέβαια και η τεχνική υποστήριξη από πλευρά των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που να εξασφαλιστεί η πλήρη συνοχή ε, μεταξύ των ευθυνών αφενό που έχουν αναλάβει αυτέ οι αρχέ και των καθηκόντων που έχουν να επιτελέσουν. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, είναι απαραίτητο τώρα νομίζω οι διαδικασίες διορισμού, ορισμού μάλλον υποψηφιωτήτων και επικύρωση των επικεφαλής αυτών των οργάνων να ολοκληρωθεί για να ξεκινήσουν τη δουλειά τους. Κάθε μέρα βλέπουμε την ε, σαφή απόδειξη της χρησιμότητας αυτών των υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά και αναφέρομαι σε διάφορα θέματα που μας απασχολούν καθημερινά στο έργο μας. Επίσης, θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω την αρχή για την αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων που θα πρέπει να αναλάβει πλήρη καθήκοντα αμέσω και είναι δική μας ευθύνη ο καθένας από, το, από την πλευρά του, από το δικό του μετερίζει να ε, συμβάλλουμε στην πλήρη λειτουργία με τους όρους που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτών των οργάνων. Και η Επιτροπή, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα μεριμνήσει έτσι ώστε να γίνει πλήρως σεβαστή η λειτουργία αυτών των οργάνων και η αποτελεσματική τους εργασία. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα έχουμε τους ομιλητές εκ μέρους των ομάδων. Ο κύριος Γκοζές, εκ μέρους της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος των Συνδημοκρατών για δυόμιση λεπτά. Κύριε Γκοζές, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε μια νομική αλλά μια πραγματικά πολιτική συζήτηση. Συζητούμε για το μέλλον της Ευρώπης ό,τι αφορά την χρηματοοικονομική ρύθμιση. Ολοκληρώνεται ένα έργο που υλοποιήσει το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο και με τη συνεργασία της Κομισιόν. Θα είμαι σαφής. Δεν θέλουμε εδώ να διασκεδάζουμε και να κάνουμε, να ε, δείχνουμε τους μίσμα ή να κάνουμε επαναστάσει. Απλώς θέλουμε να δείξουμε ότι το πνεύμα των ε, συμφωνιών μεταξύ Συμβουλίου και κοινοβουλίου έχει γίνει σεβαστό. Δεν είναι ένα μάθημα δικαίου. Τα κείμενα είναι γνωστά. Το θέμα είναι πώ θα τεθούν σε ισχύ. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για τη σαφήνεια των προτάσεών του. Ποτέ δεν αμφισβητήσαμε την Επιτροπή ούτε ε, τα όσα υπόθηκαν από την Επίτροπο, όσα υπόθηκαν από την Επίτροπο συμφωνάβουν απόλυτα μας επιθυμεί το Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια πολιτική πράξη, δηλαδή να πούμε ότι συστήνονται αυτά τα όργανα και πρέπει να του προσδώσουμε και τα απαραίτητα μέσα να λειτουργήσουν. Ε, και νομίζω ότι δεν πρόκειται απλώ για αμφιβολίε. έχουμε υποψίε σχετικά με τον τρόπο που οι διατάξει αυτέ τέθηκαν σε εφαρμογή από ορισμένα κράτη-μέλη. Γιατί τι θέλουν να ξυλώσουν την ευρωπαϊκή εποπτεία, ε, θέλουν να εμποδίσουν ε, μια χρηματοοικονομική επιπτία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκτιμούμε ότι αν αυτόν δεν ε, ήταν ε, τέτοιο τότε στις διαπραγματεύσεις ξέρετε είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες εξαιρετική δουλειά της Βελγικής Προεδρίας και σήμερα μπορούμε να βρεθούμε ενώπιον οργάνων που στην πραγματικότητα δεν θα είχαν καμία εξουσία γιατί ουσιαστικά υποσκελίζεται το προσωπικό που έχει διοριστεί. Ε, σήμερα θα πρέπει να δώσουμε μια συγκεκριμένη απάντηση στο Κοινοβούλιο και ξέρετε πόση φιλία τρέφω για σας γιατί είμαστε ε, στην ε, ίδια ομάδα. Έτσι λοιπόν ε, θέλω να σας πω ότι το πρώτο σχέδιο κειμένου δεν αρκεί. Η απάντηση του ΕΛΚ είναι απλή. Εσείς λέτε εξ ονόματος του Συμβουλίου ότι προσυπογράφετε λέξη προξέρψη τη δήλωση που έγινε από τον Επίτροπο και μπορώ να σας πω ότι για μας αυτή θα είναι μια δήλωση ικανοποιητική. Η δήλωση του Επιτρόπου είναι ακριβής, αναφέρεται σε προβλήματα ανθρωπίνων πόρων και οικονομικών πόρων, αλλά πρέπει η δική σας επιστολή να ε, ακολουθεί την δήλωση που έγινε σήμερα από τον Επίτροπο στη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των, της Ευρωπαϊκής Φιλιστικής Μαχίας Δημοκρατών, ο κύριος Μπούλμαν. Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, τι, τι συζητούμε εδώ, γιατί είμαστε εδώ. Όπω είπε και ο κύριο Επίτροπο, συζητούμε εδώ, βρισκόμαστε εδώ επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να θεσπίσει ευρωπαϊκέ εποπτικέ αρχέ άξιε του τίτλου του. Δεν ήταν αυτό όμω στα σχέδια του Συμβουλίου ούτε των κρατών μελών. Και η Επιτροπή είχε αρχικά κάποιε εμβόλειε για το κατά πόσο θα φτάσουμε στο στόχο αυτό, κατά τη θέσπιση των εποπτικών αρχών. Και θα αντιληφθείτε, θα το αντιληφθεί το Συμβούλιο, θα υποχρεωθεί να το αντιληφθεί και η Επιτροπή και μάλλον και από τις δικές εκτιμήσεις, γιατί έχουμε κάποιες ανησυχίες. Πρόκειται για μια τοποθέτηση την οποία ε, υιοθετούν όλες οι πολιτικές ομάδες, όχι εμείς ο Σεριστές, ο εκπροσωπώ, αλλά όλες οι πολιτικές ομάδες. Δεν σκοπεύουμε να επιτρέψουμε να παιχτούν παιχνίδια εθνικά εσωτερικά στην θέσπιση ή μάλλον στους διορισμούς των προσώπων που θα αναλάβουν τα ενία αυτών των αρχών. Και εδώ ακριβώς θέλουμε να έχουμε λόγο στην επιλογή των προσώπων. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις στο όντι από καιρού καιρών οι οποίες προξενούν ανησυχία. Βλέπουμε κάποιους καταλόγους, κάποιους άλλους που είναι πολύ ασαφείς, κάποιους ε, όπου δεν είναι σαφές το αν υπάρχει, αν έχει ε, επιλεγεί κάποιος για λόγους επιλογής φίλων συγκεκριμένων. Ε, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν έχουμε καθόλου υπόψη μας, δεν έχουμε ποτέ ακούσει να γίνεται λόγος για αυτά. Και ενώ υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι, άνθρωποι που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά πολύ καλά, διαπιστώνουμε ότι είναι πρόσωπα τα οποία λόγω τη απουσίας του σχετικού κύρου που απαιτεί αυτή η θέση δεν θα είναι σε θέση από ό,τι βλέπουμε να πιέσουν ή να πείσουν τα κράτη-μέλη να προβούν σε ορισμένε ενέργειε. που θα απαιτούσε η θέση του σε μια τέτοια εποπτική αρχή να πράξουν. Εκείνη η ανησυχία μα και αυτέ οι διαδικασίε είναι που μας ε, δημιουργούν το αίσθημα του ανεκανοποιήτου και γι' αυτό ερωτούμε αν υπάρχει η δυνατότητα να ε, βλέπουμε πολύ πιο ξεκάθαρα, όπως γίνεται άλλωστε και με την Όλεφ, τις θέσεις αυτές και να αποδεικνύεται ότι αυτές οι υποπτικές αρχές λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τις θέσεις του Κοινοβουλίου, γιατί δεν το έχουν αποδείξει αυτό ακόμη. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία και για την Επιτροπή και για το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τις επιφυλάξεις του Κοινοβουλίου, να μας πούν ξεκάθαρα πώς σκοπεύουν στο μέλλον να συνεργαστούν μαζί μας, να πούν ξεκάθαρα τι είδους μεταρρυθμίσεις σκοπεύουν να προβάλλουν για την περίοδο μετά το 2013 και ξεκάθαρα επίσης να πούν εάν η δική μας γνώμη ως προς την επιλογή των προσώπων θα βαρύνει στην επιλογή αυτή. Και έτσι μπορούμε νομίζω να προχωρήσουμε γρήγορα σε μια λύση νομοθετική στην ε, Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρου στην ε, Συμμαχία των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών τη Ευρώπη, κυρία Γκουλάχ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που είστε ε, εδώ ενώπιόν μας. Ξέρουμε ότι ήταν σύντομες οι προθεσμίες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, να θέσουμε σε προοπτική τι μας κινεί. Τα κίνητρά μας είναι τα εξή ότι συλλογικά για μήνες αγωνιστήκαμε έτσι ώστε να υπάρχει ένα πριν και ένα μετά την κρίση, ε, γιατί σε αυτή την ε, εσωτερική αγορά όπου διευκολύναμε την επέκταση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αναφέρομαι στις τραπεζικές υπηρεσίες ε, και στη διασυνοριακή πτυχή των υπηρεσιών. Ε, θέτουμε κοινού κανόνες και κοινή υποπτία. Και ειλικρινά, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την υποστήριξη της Κομισιόν, είδαμε ότι γυρνούσαμε γύρω-γύρω. Υπήρχαν κράτη-μέλη που ήθελαν να ελέγχουν ε, την εποπτεία, να έχουν το τελευταίο λόγο και κανένα να μην έρχεται να χώνει τη μύτη του στι υποθέσει του. Ε, μου λέτε ότι το Συμβούλιο δεν ε, έχει αρμοδιότητα για το διορισμό. Σωστό είναι αυτονομικά αλλά ο Επίτροπος υπενθύμησε ότι αυτές ε, ε, οι υπηρεσίες, για αυτές τις υπηρεσίες θα διορίζονταν κάποιοι ε, από τα κράτη-μέλη. Πρέπει εμείς να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ανεξαρτησία τα μέτρα και βούληση να προχωρήσουμε. Φυσικά γνωρίζουμε τις ευθύνε μας. Είμαστε οι πρώτοι που επιθυμούμε να τεθούν σε λειτουργία αυτές οι αρχές, γιατί εμείς συμβάλαμε στη γέννησή τους. Δεν θέλουμε να καθυστερήσει η εργασία. Σκεφτείτε τα στρε τεστ των τραπεζών, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά θα είμαστε απαιτητικοί, ε, θα ε, δούμε λεπτομερώς όσο μας είπαν οι ΜΕΝ και οι ΔΕ και θα λάβουμε μία απόφαση βάσει της συνείδησής μας. Και ευχαριστώ τον κύριο Μπαρνιέ που έκανε πάρα πολύ καθαρές προτάσεις, σαφείς προτάσεις και θα ήθελα ε, να σας παρακαλέσω να μην επιδεικνύουμε εδώ αφέλεια γιατί διακυβεύονται πολλά. Ευχαριστώ εκ μέρους των Πρασίνων Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Ο κύριος Κίκολτ. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ πιστεύω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την πραγματική δυνατότητα εφαρμογής των δυνα... το τι τον προσφέρει το δίκαιο για ουσιαστική εποπτεία στην Ευρώπη. Και πρέπει να δούμε αν θα μπορέσουμε θεσμικά να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία προσφέρεται. Βλέπουμε διαδικαστικές ελλείψεις που σημαίνουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε κατάλογο υποψηφίων ως κοινοβούλιο δεν μας δόθηκε προκαταβολικά, είδαμε μόνο ένα αποτέλεσμα τετελεσμένο. Βλέπουμε επίσης ότι δεν υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στις επιλογές των προσώπων αυτών και έχουμε αφιβολίες και προς τις διαδικασίες και το ρόλο των κρατών μελών, κατά πόσον δηλαδή αυτά εξυπηρετούν πράγματι την ευρωπαϊκή προοπτική και το συμφέρον της Ευρώπης στην επιλογή των προσώπων αυτών. Άρα λοιπόν πρέπει να θέσουμε και μια ε, εκ των βάθρων να συζητήσει τις τη διαδικασία αυτή. Αλλά πρέπει να δούμε και το κάθε πρόσωπο χωριστά, με βάση τι τις ικανότητε και δεξιότητέ του. Εδώ λοιπόν βλέπουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Βλέπουμε καταρχά από τι ε, ακροάσει ότι ένας από τους υποψηφίους δήλωσε κατά την ακρόασή του ότι δεν πρόκειται για Ευρωπαϊκή Αρχή, αλλά για ένα, ευρωπαϊκό, για ένα διακρατικό δίκτυο ε, εποπτικών αρχών. Μετά διόρθωσε βέβαια την τοποθέτησή του και επίση ερώτηση σχετική με τα λόμπι και τη διαφάνεια σε σχέση με τι ομάδε πιέσεω. Απάντηση δεν λάβαμε. Από αυτό λοιπόν για μα εξαρτάται το αποτέλεσμα τη προφορίας. Πρέπει να λάβουμε σαφεί απαντήσει σε αυτά τα δύο ζητήματα. Ευχαριστώ εκ μέρου των Ευρωπαίων Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών, η κυρία Σουίνμπερν για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Οι συντηρητικοί μεταρρυθμιστέ χαιρετίζουν την προσπάθεια να συζητηθεί σήμερα αυτή η απόφαση εδώ στον Λουμέλη, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι κατά τη δική μα ομάδα όλοι οι υποψήφοι για την, ε, την ε, υπηρεσία αυτή θεωρούμε ότι έχουν τι δεξιότητε, τα προσόντα όλα για να μπορέσουν να επιτελέσουν το ρόλο που πρέπει και όλα αυτά τα οποία λέγονται σήμερα αφορούν καθαρά τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί ούτω ώστε να γίνει ο διορισμό του. Οπότε για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον όσον αφορά του υποψηφίου, θα πρέπει αυτό να γίνει από όσο γίνεται ευρύτερο σύνολο ατόμων, τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε εξαρτησία σκέψη, αλλά και το να είναι πολύ συλλεκτική η διεύθυνση αυτών των οργάνων. Επίση, θα πρέπει ε, να ληφθεί υπόψη το πόσο ψηλέ οι είναι αυτέ τι θέσει και για το μισθό του, ε, κριτήρια, τεχνικέ δεξιότητε και ανταγωνισμό. Αυτά όλα θα πρέπει να αποφευθούν ε, να, βαρύνουν ακόμη περισσότερο, αλλά θα πρέπει να λέμε υπόψη ότι θα έπρεπε να έχουμε κάποια διαφάνεια στον αφορά το κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι όλα αυτά που λέμε θα τα λάβετε υπόψη ή στο μέλλον. Σας ευχαριστώ κυρία Σουίνμπερν. Τελευταία ομιλία εκ μέρους των ομάδων. Η κυρία Ανδρέα είναι εκ μέρους της Ευρώπης των Ελευθεριών και Δημοκρατιών. Για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι δεν ε, υπάρχει ανάγκη για αυτές τις θέσεις των εποπτών, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν και αυτές οι ίδιες υπηρεσίες, αυτοί οι οργανισμοί. Εδώ δημιουργείται, δημιουργείται ένα άλλο επίπεδο εποπτείας ε, ε, που θα αποτελέσει βελτίωση της εφιστάμενης ε, των εφιστάμενων εποπτικών αρχών. Εγώ νομίζω ότι αν πράξουμε κάτι τέτοιο απλώς θα μπερδέψουμε την κατάσταση. Ποιος είναι υπευθύνο γιατί είναι αυτός ο κανονισμός κατάλληλος για ευρύτερο χρηματοοικονομικό για μια μεγαλύτερη περιοχή το, το, του Λονδίνου, όχι, το αμφισβητώ. Δηλαδή ε, είχαμε αγνία ε, πέρσι από όσου έπρεπε ε, να εφαρμόσουν τους κανονισμούς και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι θα κάνουν κάτι καλύτερο. Για να μην αναφέρω ότι μας παρουσίασαν μόνο έναν υποψηφίο για κάθε θέση πρόκειται για μια εντελώς δημοκρατική, ένα εντελώ μη δημοκρατικό εγχείρημα, αλλά φυσικά το ίδια διαδικασία χρησιμοποιήθηκε για το διορισμό των επιτρόπων του Προέδρου, του Συμβουλίου, ε, της Αρμοστή και τα λοιπά, της και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν, εγώ θα έλεγα να ψηφίσουμε κατά αυτών των ψηφίων και οποιονδήποτε άλλων. Ευχαριστώ. Κύριος το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω. Ήμουν όσο δυνατόν πιο σαφής και ειλικρινής. Μέτρησα κάθε μια λέξη που εκφώνησα κατά τη δήλωσή μου, την οποία άλλωστε και γραπτός θα επιβεβαιώσει επιστολή που συνυπέγραψα με τον Αντιπρόεδρο κ. Σεύκοβιτς. Για να είναι σαφή τα πράγματα. Απλώς για να δώσω απαντήσεις ε, στις παρεμβάσεις, ευχαριστώ τους κυρίες και κυρίους βουλευτές, θα ήθελα να περιοριστώ σε τρία θέματα. Εξάρτηση και κύρος των επικεφαλής, των προέδρων αυτών των αρχών. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την πλήρη στράτευση του Κοινοβουλίου, την οποία άλλωστε ποτέ δεν αφέβαλα, ε, ποτέ δεν ε, ώστε αυτές οι αρχές να παραμείνουν ιστοδυνικές ανεξάρτητες. Βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο είναι θελμένο να περασπιστεί αυτήν την ανεξαρτησία και αυτό είναι πολύ θετικό. Εάν στο μέλλον δούμε τι είδους ε, και τι όγκο καθηκόντων θα έχουν να επομιστούν αυτές οι αρχές. Έγινε νωρίτερα λόγος για, τις, ε, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή για το τεστ αντοχής βλέπουμε ότι εδώ ακριβώς θα χρειαζόμαστε αξιόπιστες και ανεξάρτητες αρχές. Αξιόπιστες. Υπογραμμίζω. Αυτό είναι το πρώτο σημείο στο οποίο θέλω να επανέλθω, να σταθώ και βεβαίως το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σε αυτό συμφωνούν και φαντάζομαι και το Συμβούλιο. Η διαδικασία, οι, οι διαδικασίες για την επιλογή των προσώπων. Δεύτερο. Θυμάμαι κυρίε και κύριοι τι συζητήσει στον τριμερή διάλογο, στου τριμερεί διαλόγου, πολλαπλέ συζητήσει, οι οποίε κατέληξαν τελικά σε συμφωνία μεταξύ των συναρμόδιων για το νομοθετικό έργο ε, θεσμικών οργάνων. Στο βαθμό που κατέστη αυτό δυνατό, υπάρχει βέβαια η ρήτρα για την επανεξέταση. Δεν έχω λόγο αυτή τη στιγμή όμως να αμφισβητώ ότι ε, δεν επελέγησαν, ε, ότι επελέγησαν καλή ε, Δεν έχω κανένα λόγο δηλαδή να κατηγορήσω χωρίς περισσότερα στοιχεία ε, για ανεπάρκεια αυτούς τους ε, υποψηφίους. Και εγώ είδα τον κατάλογο έχοντας τη δυνατότητα να συναντηθώ και με τους υποψηφίους μπόρεσα να συμφωνήσω σε έναν τελικό κατάλογο ε, με βάση τα προσόντα που απεδείχθησαν κατά τη συνάντηση αυτή, αλλά η πρώτη αρχική κατάλογη, κατάλογη 165, 175 υποψηφιότητες προέρχονταν από τα διάφορα κράτη-μέλη και ασφαλώς σε αυτούς δεν είχαμε λόγο. Άρα λοιπόν ναι υπάρχει ρήτρα επανεξέτησης που μας προσφέρει την απαραίτητη εγγύηση και ως εκ τούτου δεν έχω λόγο να αμφισβητώ την επάρκεια ε, των υποψηφίων αυτών. Και ένα τρίτο σημείο ως προς την, την αντιπροσωπευτικότητα των αρχών αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα αφιστεί κόπον ώστε να επιβεβαιώνει κάθε φορά ότι αυτές οι αρχές επιτελούν το έργο τους στο απαραίτητο επίπεδο τον απαραίτητο βαθμό και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που μας στηρίζει σε αυτό το άκρος ουσιαστικό σημείο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, η νύχτα φέρνει επίτροπο και αυγή Μητροπολίτη όπω λένε. Τέτοια ώρα δεν έχω τίποτα περισσότερο να σας πω. Το μόνο εκ μέρου όλων των επιτρόπων σας παρακαλώ να επαχρυπνήσετε κι εσείς μαζί μας ώστε αυτοί οι επικεφαλής των αρχών να βοηθήσουν στο το έργο τους να πραγματοποιηθεί ουσιαστικά και παραλαμβάνω και υπογραμμίζω δεν υποκαθιστούν τις εθνικές αρχές εποπτείας, τις συμπληρώνουν όμως το έργο τους έναντι προκλήσεων μεγάλων και κινδύνων που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε ανάγκη να έχουμε αυτά τα όργανα τα ευρωπαϊκά, αυτές τις αρχές εποπτείας που θα αποτελούν κατά κάποιο τρόπο το ραντάρ που θα εντοπίζει τους κινδύνους από όπου και αν προέρχονται Αγορέ κινούνται πολύ πιο γρήγορα από εμά, κυρίε και κύριοι, γιατί η δημοκρατία, η σύγχρονη δημοκρατία απαιτεί και λίγο χρόνο παραπάνω. Αυτή τη δουλειά όμω μπορούν αυτές οι αρχέ να την επιτελέσουν πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει εκ μέρου του Συμβουλίου κυρία Τζούρη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, πρώτα πρώτα επιτρέψτε μου να σα απαντήσω αυτή την ερώτηση η οποία τόσο συχνά α, α, ναι, ανευθύ σε αυτή την ερώτηση γιατί όσον αφορά τους κανονισμούς γιατί ξέρουμε ότι η ίδια η τυρλική παράγραφος είναι εκείνη η οποία λέει ότι όσον αφορά τους ορισμούς και διορισμούς των Προέδρων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά τα οποία έχει υποβάλει ως προτάσεις οργανισμών επίσης το άρθρο 89 των κανονισμών επίσης προβλέπει να γίνει μια αναθεώρηση από την Κομισιόν προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 2014 και κάθε τρία χρόνια. Επομένως με αυτή την ε, διάταξη πρόκειται εν αυτό το χρόνο να αναθεωρήσουμε αυτόν τον κανονισμό λαμβάνοντα υπόψη την ε, πρακτική εμπειρία και έτσι θα έχουμε υποδομητικό διάλογο των θεσμικών οργάνων και έτσι θα στώσουν τον δρόμο για τις μελλοντικές εξελίξεις στα Ουγγρικά. Στην μερική μου γλώσσα, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, θέλω να σα πω ότι δεν υπάρχει κανένα είδου ε, διαφωνία μεταξύ ημών και ημών όσον αφορά την ουσία αυτών των θεμάτων και όλοι ενδιαφερόμεθα ούτω ώστε να υπάρχει μια ισχυρότερη Ευρώπη και να έχει ισχυρά θεσμικά όργανα. Και αυτό αφορά και την χρηματοπιστωτική εποπτεία. Και εμεί ε, έχουμε επιτελέσει έργο δύσκολο εσείς και εμείς το Συμβούλιο. Αυτό έγινε ως αποτέλεσμα αυτής μας προσπάθειας οπότε και τα θεσμικά όργανα θα είναι έτοιμα ούτως ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής μετά την κρίση και να παρασχεθούν οι εγγυήσεις που πρέπει για να λειτουργήσουν εύρεθμα οι αγορές ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να θρακιστεί το ευρώ. Πάντως δεν υπάρχουμε ούτε προστριβή και διαφωνία εσείς και εμείς όσον αφορά το πώς θα πλαισιωθούν αυτά τα νέα όργανα, αυτές οι νέες υπηρεσίες. Σας ανέφερα ποιες είναι οι κείμενε διατάξει που θυμίζουν αυτού του ορισμού και διορισμούς και συμφωνώ μαζί σα ότι θα πρέπει αυτέ οι αρχέ να διέπονται από πολιτική διοίκηση. Δεν θα πρέπει να είναι απλά η επέκταση των εθνικών ε, ομολόγων του. Θα πρέπει να είναι αυθεντικά ευρωπαϊκέ υπηρεσίε. Εγώ στην ε, εισήγησή μου επικεντρώθηκα στις αρμοδιότητες αυτών των υπηρεσιών. Έχουμε επίσης λάβει και την επιστολή του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής και ε, εγώ ασχολήθηκα με τα όσα έχουν σχέση με το δικό μου χαρτοφυλάκιο οπότε και τονίστηκαν το τι εγγύσεις υπάρχουν τόσο να λειτουργούν ανεξάρτητα αυτές οι υπηρεσίες. Και επίσης ως συνομοθέτης για τον ε, προπολογισμό θα πρέπει να σας εξασφαλίσω ότι θα υπάρξει εύρυθμη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά τους και έτσι με όλες αυτές τις υπηρεσίες θα έχουμε ελπίζω καλύτερε επιτές στο μέλλον ο δε προεδρεύων του ΕΚΟΦΗΝ απήντησε στον πρόεδρο της Οικονομικής σας Επιτροπής με επιστολή τη δε απάντηση αυτή ελπίζω να την κρίνετε ικανοποιητική. Έχουμε αυτή την γλυκά ε, εναλλασσομένη προεδρία κύριε Γκοζές και αυτή η προεδρία σύμφωνη με τις θέσεις αυτές που είπατε. Δεν νομίζω να υπάρξει κανένα είδους πρόβλημα. Όσον αφορά την επιλογή διορισμού αυτών των υποψηφίων. Ευχαριστώ πολύ και τώρα στην για διάταξη έχουμε την κοινή συζήτηση για το θέμα της μπανάνας. Έχουμε καταρχάς μια σύσταση κυρίας Μπαρτζάνη.